θέση του Συμβουλίου. Δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού μας ε, θα υπογράψει την απόφαση αυτή ο Πρόεδρος. Αποκινούμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μέσα στο μεσημέρι σήμερα. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μορέιρα. Έλεγχο εξαγωγών μεταφορά μεσητείας διαμετακόμιση ειδών διπλής χρήσης. Δεν υπάρχει πρόταση απόρριψη ούτε κάποια τροπολογία. Επομένως κηρύσω εγκριθήσα την θέση του Συμβουλίου και περνάμε στην ψηφορία της εκθέσεως Λάγκεν για τα παράγωγα και να δώσω το λόγο καταρχάς στον Επίτροπο, στον Επίτροπο κ. Ταγιάννη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της συμφωνίας για το ΕΜΙΡ, αλλά έχει κάποιες επιφυλάξεις νομικές σχετικά με το άρθρο 67 παράγραφος 3. Θεωρεί ότι το άρθρο αυτό πρέπει να διαγραφεί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άρθρο 290 θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εξής είναι κάτι το αυτόνομο σχετικά με την προπαρασκευή και την έκδοση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Οι συνέπειες στις συμφωνίες που έχουν ήδη υπάρξει ανάμεσα στα τρία όργανα αντικατοπτρίζουν άλλωστε αυτού του είδους την ερμηνεία. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι απαράδεκτο και αντίθετο με το γράμμα και πνεύμα του 290 να ξεπεράσουμε τα όρια της αιτιολογικής σκέψης που προβλέπεται από το πρωτόκολλο και να μην υπάρξει υλική εφαρμογή διαφορετική από αυτήν που έχει ήδη υπάρξει. Κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για αυτό το νομικό θέμα θα τοποθετηθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο απέριψαν το αίτημα της Κομισιόν και τα δύο νομοθετικά σώματα λοιπόν συμφωνούν θα ήθελα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ορισμένα πράγματα για το έργο αυτό. Εγκρίνουμε με τον ε, κανονισμό αυτόν ένα βασικό κομμάτι της ρύθμισης των ε, χρηματαγορών. 3,5 χρόνια μετά τη χρεοκοπία της ε, Λίμαν διασφαλίζουμε πως παράγωγα εκτός χρηματιστηρίων θα πρέπει να δηλώνονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο και να καλύπτονται με ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για 708 τρισεκατομμύρια ε, ε, δολάρια ΙΠΑ. Μιλάμε για πολλαπλάσιο του παγκοσμίου ΑΕΠ. Επιτέλους λοιπόν μπαίνει μια τάξη σε αυτή την τεράστια και αδιαφανή αγορά. Θα υπάρχουν κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι και αποθετήρια τα οποία θα πρέπει να εμπλέκονται σε κάθε συναλλαγή και θα υπάρχει και ρύθμιση θε... χρηματοπιστωτικών δρυμάτων τρίτων κρατών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους και την Κομισιόν, τον κύριο Μπαρνιέ. Λυπηρό θεωρώ το ότι ο κανονισμός για μια τόσο σημαντική ψηφοφορία δεν μας επιτρέπει συζήτηση. Δεδομένου λοιπόν του λεγόμενου τριμερούς ε, ατύπου διαλόγου ζητάω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί Ιούλιο του 2012 θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί αυτό το θέμα και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Κυρία Μπόουλ, ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώνω αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν για το άρθρο 67.3. Αλλά δεν σκοπεύουμε να το διαγράψουμε. Το άρθρο λέει πριν υιοθετηθεί μια πράξη κατεξιοδότηση, η Κομισιόν θα προσπαθήσει να συμβουλευτεί την ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ δεν είναι ειδική των κρατών μελών, είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και εμείς υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία της αρχής αυτής. Δεν είναι ειδική των κρατών μελών, ούτε επιβάλλεται μία υποχρέωση με αυτό. Γι' αυτό το λόγο και για άλλους δεν συμφωνούμε με την άποψη της Κομισιόν πως παραβιάζει το άρθρο 290 της Συνθήκης της Ένωσης, ούτε τη Διοργανική Συμφωνία, την οποία επίσης ανέφεραν. Και θέλω αυτό να γραφτεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπόλς. Θέτω σε ψηφορία λοιπόν την έκθεση Λάγγεν ξεκινώντας με την τροπολογία 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία ψήφο εκεί στο βάθο. Εγκρίνεται λοιπόν τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψήφισματο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Μωρέ Σαχτιέ. Ελάχιστε απαιτήσει υγεία και ασφάλεια όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων συγκίνητων περιεχόμενου. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται την πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση νομοθετική υπέρ μάλλον το, το νομοθετικό ψήφισμα ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση ΚΑΖΑ, Διοικητική Συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωση. Οι τροπολογίε 12 και 14 δεν αφορούν όλε τι γλώσσε, άρα δεν θα τι θέσω σε ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφο 1, εδάφιο Δέλτα του κανονισμού, θα αναζητήσουμε την κατάλληλη γλωσσική λύση με του ενδιαφερομένου. Έκθεση τώρα, πρόταση κανονισμού ουσιαστικά Μία δέσμη τροπολογιών 2 έως 11, 13, 15, 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται οι τροπολογίες αυτές. Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητή. Μάλλον όχι. Θα ψηφίσουμε την πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και το ψήφισμα μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση ΒΟΝ προβλέψει εσόδων και δαπανών για το 2013. Πριν ένα κοινοβούλιο. Ξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματο και ξεκινούμε με το αρχικό κείμενο τη παραγράφου 2, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 ονομαστικά ψήφι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστικά και αυτή. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε συνολικά τώρα το σχέδιο του ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Le vote pas alors... Δεν είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, είπα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη έκθεση, έκθεση Ματέρα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η τροπολογία 2, ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα ονομαστικά το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση Λαμασούρ. Τροποποίηση του κανονισμού υπό το φω εξέλιξη των σχέσεων με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τι εθνικέ κυβερνήσει. Τροπολογίες 1 έως 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα το, την πρόταση συνολικά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριο Λαμασού. Υπάρχει έτοιμα επί της διαδικασίας για τον κύριο, από τον κύριο Μικάλσκι πριν ψηφίσουμε για τη Λευκορωσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όπως θα θυμάστε πριν από δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την ε, κατάσταση στη Λευκορωσία ε, κατά δύο εβδομάδες ε, για μία μέρα Μάλιστα μετά την ε, άρνηση από τον κύριο Λουκασέγκα να δώσει χάρη σε άτομα τα οποία είχαν καταδικαστεί για τις επιθέσεις ε, στο Μίνσκ. Είχα πει τότε πως ε, θα το ερμήνευαν ως ένα μήνυμα αδυναμίας και δυστυχώς είχα δίκιο. Οι δύο αυτοί νέοι εκτελέστηκαν την επόμενη μέρα. Και αυτό τονίζει αυτό το οποίο πάντα λέω, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Λευκορωσία και τον κύριο Λουκασάνκα. Και ελπίζω να μην ε, κάνουμε πίσω στις ε, προσπάθειές μας ε, για να φροντίσουμε οι άνθρωποι στη Λευκορωσία να ζουν με αξιοπρέπεια. Σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε το ψήφισμα. euh... Ah, Monsieur la parole également. Κύριε Ποτασέβη, θέλετε και εσείς το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μιγκάλσκι. Πράγματι, και εγώ σας ε, καλώ να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα και όλες τις τροπολογίες, αλλά δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση του κυρίου Μιγκάλσκι. Δεν συμφωνώ πως ήταν αδυναμία από μέρους μας και αυτή οδήγησε στις εκτελέσεις. Οι εκτελέσεις πιθανότατα έλαβαν χώρα πριν από την απόφασή μας. Στην αρχή της ε, εβδομάδας του Στρασβούργου το κράτησαν μυστικό στη Λευκορωσία. Δεν ξέρουμε πότε εκτελέστηκαν ακριβώς. Οπότε νομίζω παραπάει να λέμε πως η απόφασή μας οδήγησε στην επιδείνωση της κατάστασης. Ελπίζαμε πριν από δύο εβδομάδες σε αλλαγή στην πολιτική της Λευκορωσίας. Δυστυχώς δεν επιτύχαμε και σήμερα πραγματικά δεν υπάρχει, δεν νομίζω, δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με όσους συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Ο κύριο Βίγκενιν έχει χτίσει το λόγο. Διαδικαστικό λέει ο κύριο Βίγκενιν. Διαδικαστικό. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Εγώ υποστηρίζω αυτά που είπε ο κ. Πρωτοσέβιτς, αλλά χθε το απόγευμα την τελευταία στιγμή ζητήθηκε από τους συντηρητικούς να υπάρξει καταδιέρεση ψήφος στο 6 και στο 2. Η σοσιαλιστική ομάδα δεν μπόρεσε να αντιδράσει, θα ήθελα όμως να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα της θανατικής ποινής και πρέπει για μια ακόμη φορά να ζητήσουμε την κατάργησή της. Θέλουμε αυτό να γίνει με ξεκάθαρο αποφασιστικό και διαφανή τρόπο. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την ονομαστική ψήφο. Ναι, έχω αντίρρηση να υπάρξει ονομαστική ψήφος. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Υπάρχει ξεκάθαρη διαδικασία όταν ζητείτε και όταν κάποιοι θέλουν να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία πρέπει να ακολουθούν την ορθή οδό. Γιατί ξαφνικά αν κάποιος ζητάει να υπάρξει ονομαστική ψήφο, ο καθένας προς το συμφέρον του μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν 40 οι οποίοι να συμφωνούν με τον κύριο Πάτεν για την απόρριψη του αιτήματο Βίγγενιν. Συνεπώς το αίτημα για ονομαστική ψήφο γίνεται δεκτό και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. On compte, on compte. Oui, ça. C'est plus ou moins 40. Bien. Sans en avoir la totale certitude, je pense qu'il y a 40 personnes qui se sont levées. Νομίζω ότι έχουν ήρθει ε, 40 ε, βουλευτέ, οπότε δεν θα γίνει ε, δεκτό το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Donc on euh, Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα, τροπολογία 6, σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό Τέσσερα. υπέρ κατά αποχές δεκτό Πέντε υπέρ κατά αποχές δεκτό το ψήφισμα ως έχει ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή περνάμε τώρα στις προτάσεις ορισμού των μελών της ειδική Επιτροπής για την Διεθνή Εγκληματικότητα. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στις προτινόμενες υποψηφιότητε θεωρούνται δεκτές. Περνάμε τώρα στον κύριο Λάμστορ στην έκθεσή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Δεκτή η πρόταση Λάμστορφ. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματο για την διεύρυνση ε, σχετικά με τη Σερβία. Ο κύριο Κάτσιν, Κατσίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρατήρησα πως η Σερβία δεν έχει στείλει ακόμα υπογεγραμμένη συμφωνία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στον μεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Πριστίνα, τον κύριο Ρόμπερτ Κούπερ, η οποία υπογράφηκε στις 15 ε, Φεβρουαρίου στην ε, Πριστίνα. Γι' αυτό έγινε και υποψήφια χώρα η Σερβία. Η Πριστίνα απέστειλε το επίσημο υπογεγραμμένο αντίγραφο, ενώ το Βελιγράδι δεν το έχει ακόμα κάνει. Η εφαρμογή της Συμφωνίας Διαχείρισης των Συνόρων είναι εξαιρετική σημασία. Καλό την σερβική κυβέρνηση να υποβάλει αυτό το έγγραφο και να διατηρήσει άρα την αξιοπιστία της και να επιδείξει την δέσμευσή της για την εφαρμογή της συμφωνίας. Μιλώ εξ ονόματος όλων των σχεδόν εισηγητών, τους οποίους ευχαριστώ για το επικοδομητικό τους έργο στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Κατσίν. Περνάμε στις φοφορίες. Ξεκινάμε με το απολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 6 έχει καταπέσει. Η 4 τώρα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 7 έχει καταπέσει, περνάμε στην 8, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 5, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τοπολογία 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές δεκτή. Το ψήφισμα στο σύνολό του, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Τέλος. Ε, συγχαρητήρια δεκτή. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος για τη διεύρυνση σχετικά με το κοσυφοπέδιο. Η κυρία Λούνατσεκ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους πιο για την επικοδομητική συνεργασία στην ε, έκθεσή μας η οποία υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική του πεδίου. Έχω μία παρατήρηση και ένα αίτημα. Η παρατήρηση είναι πως από όταν ψηφίστηκε η έκθεση στην Επιτροπή εξωτερικών πέρασαν δύο μήνες. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο. Έκτοτε έχουν συμβεί πολλά πράγματα μέσα και γύρω από το Κοσμοπέδιο, π.χ. το θετική κατάληξη των συνομιλιών με το Βελιγράδι και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που άνοιξαν το δρόμο για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του Κοσμοπεδίου. Γι' αυτό κατέθεσα οι ίδια 11 τροπολογίες που αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα. Να σα ζητήσω λοιπόν να τη στηρίξετε. Ένα αίτημα προς τους ε, σοσιαλδημοκράτες για την πρώτη τροπολογία που θα ψηφίσουμε τώρα, την υπαριθμών 13 και αφορά τον, την έκβαση του διαλόγου. Θεωρώ πως το να μπει αυτή η τροπολογία στην αρχή δεν είναι κάτι το σωστό. Πρέπει να πάει στην παράγραφο 2 που αναφέρεται στο διάλογο και θέλω να ζητήσω από τον εισηγητή και την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών να δεχτούν ε, να πάει αυτό το αυτή η τροπολογία σε άλλο μέρος. Αν δεν το δεχτούν οι σοσιαλδημοκράτε, ζητάω από τους συναδέλφου να την καταψηφίσουν, γιατί τα ζητήματα αυτά καλύπτονται στην παραγραφό 2. Ευχαριστώ. Κύριε Ρούτσακ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε κατά του να αλλάξει θέση. Θέλουμε να γίνει ψηφοφορία με το κείμενο ως έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Check à savoir si oui ou non. On le laisse tel quel Ok. Ok. Εντάξει, θα απορριφθεί επομένω από τα τη κυρία Λούνατσα και ψηφίζουμε την τροπολογία 13 υπέρ. Και contre. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 13 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est fermé. Κατά. Τέλος της ψηφοφορίας μάλλον. Απορρίπτεται. Η 14 τώρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψήφος. Πέρα τη ψηφοφορίας. Δεκτή. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία μάλλον. Τέλος. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τοπολογία 3. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία της κυρίας Λούνατσεκ. Ποιοι είναι υπέρ. Α, για μια στιγμή. Η κυρία Λούνατσεκ το αποσύρει. Έχετε το λόγο κυρία Λούνατσεκ. Νόμιζα πως ε, επειδή είναι στο κείμενο η τροπολογία δεν χρειάζεται να την αναφέρω. Μιλάει για τα επίκαιρα γεγονότα των τελευταίων δύο-τριών ημερών για να μπουν στην έκθεση. Η τροπολογία λοιπόν πρέπει να έχει ως εξής. Καλωσορίζει την πρόθεση της Κομισιόν να κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας για συμφωνία σύνδεσης Κοσφοπεδίου Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως σημειώνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Δευτέρου του 12 και καλωσορίζει ιδιαίτερο στην ε, επίσημη έναρξη αυτής μελέτης από τον Επίτροπο Φίλη την 25η Μαρτίου κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί το αργότερο, το φθινόπωρο του 12. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις σε αυτήν την προφορική τροπολογία. Όχι, την ψηφίζουμε λοιπόν. Α, υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τοπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τοπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 για μια στιγμή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 8 ψηφίζεται πέρα της φοφορίας υπέρ ζητώ συγγνώμη γίνεται δεκτή Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές είπα. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Για την 10 ψηφίζεται. Πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τοπολογία 11 τώρα ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο στο σύνολό του, ονομαστική ψήφος. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Έχουμε την 17, ποιοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην 26 υπάρχει προφορική τροπολογία της κυρίας Όμερ Ρόιτεν. Έχει κάποιος κάποια αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Μπορείτε να την παρουσιάσετε. Κυρία Όμεν Ρόιτεν, πού είστε. Θα ήθελα να προσθέσω ως προφορική τροπολογία ε, εθνοτικές και θρησκευτικέ κοινότητες.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 θα αναγνώσω το κείμενο της προφορικής ε, τροπολογίας για την κατάσταση της ε, τροπολογίας 14 καταδικάζει στην άρα τις πρόσφατες επιθέσεις ε, κατά ευρωπαϊκών γραφείων, τουρκικών εφημερίδων και ζητά να υπάρξει συντονισμένη έρευνα των επιθέσεων αυτών. Voilà. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς είχαμε καταθέσει την αρχική τροπολογία, λυπούμεθα για το ότι δεν ε, υπήρχε δυνατότητα να αφαιρθεί η εφημερίδα Ζαμάν γιατί ήταν τα γραφεία αυτής της εφημερίδας που χτυπήθηκαν σε Παρίσι, Λονδίνο, Ζηρίχη και Ρότερνταμ. Αλλά παρόλα αυτά θα υποστηρίξουμε την ε, τροπολογία γιατί είναι βασικό στόχος η ελευθερία του τύπου. No. Ποιοι είναι κατά αυτής της φοφορική τροπολογίας. Μπορεί να ψηφιστεί λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ της 14. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οι 5 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 19. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη στις ψηφοφορίες Απορρίπτεται. Οι τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 39 τώρα. Το πρώτο τμήμα ονομαστική ψήφος. Πέρα της ψηφοφορίες. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα ονομαστική ψήφος. Πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτό. Τροπολογία 15. Ονομαστική ψήφος επίσης ψηφίζεται. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 20 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 48. Το αρχικό κείμενο ονομαστική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 27 τώρα, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 50. Κραυκικό κείμενο πρώτα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ξανά ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Δεκτό. Η επτά ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η οκτώ ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι προφανές. Τίθεται σε ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο λοιπόν. Η οκτώ ψηφίζεται. Απορρίπτεται. Η εννέα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Ονομαστική ψηφοφορία για την 22. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η δέκα υπέρ κατά δεκτό 58 έχω εδώ μία προφορική τροπολογία του κυρίου Ντάτμουθ κύριε Ντάτμουθ έχετε το λόγο χωρίς μικρόφωνο κύριος Ντάτμουθ Mettez votre micro, il n'est pas allumé. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα αναφέρω την προφορική τροπολογία. Θεωρεί πως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία θα πρέπει να ανασταλούν μέχρι η Τουρκία να καταργήσει τη συμφωνία κατάργησης βίζας που υπέγραψε το 2009 με το καθεστώς του Προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Ασάντ amendement oral. Προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Α, υπάρχει μία αντίρρηση. Bien, donc cet amendement oral n'est pas retenu puisqu'il y a plus de 40 personnes. Madame, comment s'appelle là Madame Omen Reuten, vous voulez la parole Je vous la. Κυρία Omen Reuten, έχετε le λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Όμεν Ρόιτεν, ησυχία. Κυρία Πρόεδρε, αυτό δεν έχει σχέση με προφορική αλλαγή του κειμένου. Είναι μια κανονική τροπολογία που έπρεπε να έχει σαχθεί στην κανονική διαδικασία. Είμαι κατά. Euh, Περνάμε στην τελική ψήφο τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε, τώρα. στην ψηφοφορία για την ε, έκθεση για τη διεύνηση ό,τι αφορά το Μαυροβούνιο. Ναι. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε στην έκθεση Μπόντου, πλαίσιο εταιρική διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κύριε Μπόντου, έχετε προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 1. Έχετε το λόγο. Allumez votre micro. Okay. Mulțumesc. Aș dori să adaug cuvântul voluntar la punctul... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθεθεί στο 11α, ε, συγγνώμη 18, ε, η λέξη voluntary, volunteer, εθελοντικό. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία με αυτή την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 3. Εντάξει, θέλετε να ελέγξουμε. Ευχαρίστως. Ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Δεν είναι προφανές. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μποντού. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ιβάνοβα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τροπολογία 1. Ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 39. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 80. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 81. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 89 ε, κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ σκόντε τα χέρια σας. Παράγραφος 95 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 114 τώρα, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του ψήφιντος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κύριε Γκέμπελς. Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πήγατε λίγο γρήγορα σε ό,τι αφορά την ψήφιση του δεύτερου τμήματος ε, της τροπολογίας 89. Θα παρακαλούσα ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Λυπούμε, λέει πρόεδρος, αλλά εγκρίθηκε και δεν μπορώ να ικανοποιήσω το έτοιμά σας. Τελική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Βαλεάν. Έκθεση 2010 για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 1 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 30 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αμφίροπο το αποτέλεσμα. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Είδατε. Εγκρίνεται μένα, αλλά με δύο ψήφους διαφορά μόνο. Πού είμαστε τώρα. Α, στην αιτιολογική σκέψη. Άι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα συνολικά το ψήφισμα τάσω στη χειρός, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Και Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Κύριε Λάμσδορφ, έχετε το Παρακαλώ, ησυχία. Στον κατάρογο των ε, ψηφοφοριών η έκθεσή μου περιγράφεται ως έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, αλλά πρόκειται για μια σύσταση προς το Συμβούλιο. Διαφορετικός χαρακτήρας. Δεν έπρεπε να το έχουμε ψηφίσει καν σύμφωνα με τον κανονισμό και αν υιοθετηθεί δεν πρέπει να ε, γίνουν δεκτές οι τροπολογίε των ομάδων. Παρακαλώ λοιπόν να διορθώσετε αναλόγως τα έγγραφα. Μάλιστα κύριε Λάμσδορφ. Θα το λάβουμε υπόψη μας. Περνούμε λοιπόν σε αιτιολογήσεις ψήφου.